Mesdames, Messieurs, Ξεκινάμε τις εργασίες μας. Δεν έχουν έλθει όλοι οι συνάδελφοι, ιδιαίτερα από τις δύο πανίσχυρες ομάδες, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και το Σοσιαλιστικό που εκπροσωπούνται από εκλεκτούς μεν συναδέλφους αλλά ολίγους δε. Ελπίζω να έρθουν σύντομα. Έχετε λοιπόν μπροστά σας την ημερήσια διάταξη. Θα πρέπει εδώ να αναφέρω ότι η παρουσίαση της μελέτης πώς ε, χρησιμοποιούν τις συνεισφορές στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό αναβάλλεται. Ε? Ναι. Οι ψηφοφορίες θα ξεκινήσουν αύριο την 9η πρωινή και αμέσως μετά στις 10 θα ξεκινήσουμε την ακρόαση για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Θα πρέπει να ψηφίσουμε για τα δύο θέματα τα οποία αφορούν το δημοσιονομικό κανονισμό, επί του οποίου υπήρξε τελικά μια συμφωνία στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας με τους εκπροσώπους του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ε, συγχαίρω εδώ τον εισηγητή μας. Ε, θα πρέπει κανονικά να έχουμε μια συνεδρίαση που θα τελειώσει νωρίς σήμερα, κάτι το οποίο θα μας επιτρέψει αμέσως μετά να οργανώσουμε τους συντονιστές εποφελούμενοι της παρουσίας των διερμηνέων, όσων διερμηνέων χρειαστούμε. Ε, το λέω αυτό ήδη έτσι ώστε οι συνεργάτες ήδη να ειδοποιήσουν τους συντονιστές για να είναι παρόντες σύντομα εδώ. Δεν υπάρχουν λοιπόν παρατηρήσεις για την ημερήσια διάταξη, θεωρείται δεκτή. Οι ανακοινώσεις του Προέδρου πλέον αφορούν το κομπουνιούζ, είναι στο κομπουνιούζ και σας προτείνουν λοιπόν αμέσως Σχετικά με το σημείο 3, καταρχάς την έγκριση των πρακτικών των προηγούμενων συνεδριάσεων. Έχει διανεμηθεί η συνεδρίαση της 19ης Μαρτίου και αν δεν υπάρξουν ως συνήθως παρατηρήσεις μέχρι το τέλος της συνεδρίασης θεωρούνται τα πρακτικά αυτά δεκτά. Ε, περνάμε λοιπόν άμεσα στο σημείο 4 η ομάδα παρακολούθησης των εργασιών της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και ιδιαίτερα στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Ενθυμίστε ότι μετά από το αίτημα των ισογητών μας για τον προϋπολογισμό του 14 και του 15, η Γένσεν και Γαρδιά Σαβάλ, οργανώσαμε εμείς μια συζήτηση με τον Επίτροπο Λεβαντόφσκι και την Επίτροπο Γεωργίευα στις 4 Μαρτίου. Πήραμε συμπληρωματικές πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα της ανθρωπιστικής κυρίως βοήθειας και οι δύο εισηγητές, χάρη ακριβώς στις πληροφορίες οι οποίες τους δόθηκαν εκείνη τη στιγμή και από τότε, α, θέλησαν να έχουμε την δυνατότητα σήμερα να συζητήσουμε, να οργανώσουμε μια ανταλλαγή απόψεων γύρω από το Monitoring Group με τους υπευθύνους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που, ακολουθούν, που παρακολουθούν τα θέματα των πιστώσεων πληρωμών στην ανθρωπιστική βοήθεια γενικά και γενικότερα σε θέματα εξωτερικής δράσης. Ακόμα και αν όπως ακριβώς και ο Γενικός, Γραμματέας, ο Γενικός Διευθυντής Προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα μας υπενθυμίσει, τα προβλήματα των πιστώσεων πληρωμών αφορούν το σύνολο των γραμμών του προϋπολογισμού και όχι μόνο αυτά στα οποία θα αναφερθούμε σήμερα. Έχουμε λοιπόν ανάμεσά μας και τους ευχαριστώ για αυτό ε, τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, εξ ονόματος της Γενικής Διεύθυνσης Προϋπολογισμού, τους ομολόγους μας, ε, συνομιλητές μας, από την Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ, τον Γενικό Διευθυντή Σόρεντσεν και τον κύριο Μπρούνερ που είναι Διευθυντής για τους ιδίους πόρους και τις εταιρικές σχέσεις, όπως και τον κύριο Μάρκο Πανιγκάλη, τμήματάρχη και από την ΤΕΦΚΟ έχουμε τον κύριο Λουκ Μπαγκούρ, ο οποίος είναι Διευθυντής ε, ε, Διαβέσιμων Πόρων και τον Μίκαελ Κέλλερ, ο οποίος με τη σειρά του είναι υπεύθυνος για τα θέματα γειτονίας. Και τον κύριο Μάργκε, αν ακούσαμε καλά το όνομα, ο οποίος είναι α, διευθυντής για τα μέσα εξωτερικής πολιτικής. Λοιπόν, ο εισηγητής θα ήθελε το λόγο για να κάνει μια εισαγωγή στη συζήτηση, η κυρία Γένσεν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι αρχικά θα έλεγε κανείς ότι με την συζήτηση την οποία είχαμε με την κυρία Γεωργίευα και με τον Επίστροπο Λεβαντόφσκι ε, το θέμα αυτό το ξεπεράσαμε. Νομίζω όμως ότι υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία είναι σε εκκρεμότητα και δεν μπορούμε εμείς ε, παρά να υπογραμμίσουμε όσο περισσότερο γίνεται το θέμα αυτό. Όλοι συμφωνούμε σε πολιτικό επίπεδο ότι η ανθρωπιστική βοήθεια δεν πρέπει να πέσει θύμα της έλλειψης πόρων και δυστυχώς αυτό συμβαίνει. Συγγνώμη. Είναι ένα θέμα λοιπόν το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε άμεσα. Η κατάληξη δεν ήταν αυτή που περιμέναμε. Έχουμε θέσει αρκετές ερωτήσεις, τις οποίες έχετε ήδη στην διάθεσή σας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εμβαθύνουμε επί της ουσίας για το πώς οι καθυστερήσεις πληρωμών έχουν αρχίσει να σωρεύονται. Είδαμε εμείς να υπάρχει μεγάλη αύξηση των ανακών στην ανθρωπιστική βοήθεια ε, επίση και μια αύξηση στις υποχρεώσεις, αλλά διαπιστώνουμε όμως ότι η ικανότητα πληρωμής είναι ιδιαίτερος περιορισμένη και περιορίζει σαφώς αυτά τα οποία μπορούμε να πράξουμε και δεν αντιστοιχεί με τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πήραμε λοιπόν τις απαντήσεις στις ερωτήσεις μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για τις απαντήσεις αυτούς που τις έστειλαν, διότι εμβαθύνουν στο θέμα, το διαφωτίζουν και μας διαφωτίζουν. Στην ουσία εμείς σπρώχνουμε και μεγαλώνουμε μια τεράστια χιονόμπαλα η οποία αντιπροσωπεύει την αύξηση των ε, υποχρεώσεων που δεν μπορούμε να τιμήσουμε και δεν μπορούμε να αναλάβουμε και νέες πρωτοβουλίες γιατί δεν έχουμε πλέον την ικανότητα να τις πληρώνουμε. Υπήρξαν και κάποιες άλλες επιπλέον πληροφορίες στο υλικό το οποίο λάβαμε. Το θέμα του τόκου, διότι εμείς καθυστερούμε την πληρωμή της ΜΚΙΟ και ταυτόχρονα ε, τα επιτόκια ε, για τις οργανώσεις αυτές αρχίσουν να είναι ιδιαίτερα υψηλά, ιδιαίτερα σχετικά με τα ποσά τα οποία χρειάζεται να πληρώσουμε. Ε, τώρα το 2013 μιλάμε για 300 σχεδόν χιλιάδες ευρώ και δεν έχουμε χρήματα. Ο προϋπολογισμός μας είναι μικρός και είναι χαζό να χάνουμε τα χρήματά μας ακριβώς επειδή δεν τα έχουμε ή δεν έχουμε όσα θέλαμε. Λοιπόν, θα ήθελα να ακούσω τις παρουσιάσεις τις οποίες θα κάνουν οι κύριοι κύριοι Σόρενσεν και οι συνάδελφοί του για να καταλάβουν οι συνάδελφοι καλύτερα το τι σημαίνει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τα υλικά τα οποία μας απέστειλαν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κατανοήσει κανείς τη σοβαρότητα της κατάστασης. Το θέμα δεν είναι αυστηρά τεχνικό. Το θέμα είναι πραγματικά ουσιαστικής μείωσης της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ανθρωπιστικής πολιτικής. Και εμείς θέλουμε να κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Υπάρχει μια ηλυμένη πολιτική απόφαση και αυτό αυτή η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Επιστρέφω λοιπόν το λόγο σε εσά κύριε Πρόεδρε για να συνεχίσετε τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Αν ο κύριος Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να υπενθυμίσω κάποια δεδομένα, βασικά στοιχεία, σε σχέση με την κατάσταση των παρελθόν και τον τρόπο με τον οποίο εμεί, ω Γενική Διευθυνσία του Προπολογισμού, απολογίζουμε να διαχειριστούμε την κατάσταση του επόμενου μήνε. Οι συνάδελφοι θα επισέλθουν σε τι λεπτομέρειε σε σχέση με τον κάθε τομέα αρμοδιότητά του. Θα ήθελα λοιπόν να υπενθυμίσω πρώτον ότι για το 2013 η εκτέλεση του προπολογισμού έφτασε επίπεδα ανευπροηγουμένου και στις δεσμές οχρώσεων και στις πληρωμές και παρά, σημειώνω, τις σημαντικές αυξήσεις που σημειώθηκαν από την αρχή του έτους, τα 11 δις που είχαμε, τα 11,8 δις που είχαμε να κάνουμε, που είχαμε επιπλέον στον προπολογισμό. 11,2 ε, δις, συγγνώμη. Και έχουμε να κάνουμε με μία μείωση τα 4,5 δις ε, στον τομέα της συνοχής, αντίστοιχη αύξηση στους υπόλοιπους ε, τομείς. Στο κεφάλαιο 4 η κατάσταση πάλι παραμένει συνεπής με τα όσα λέω τώρα, γενικά για τον προπολογισμό. με απορρόφηση σχεδόν 100%. Χρήση για τις ε, δεσμεύσεις υποχρώσεων αλλά και απορρόφηση για τις πληρωμές και αυτό παρά την αύξηση κατά 500 εκατομμύρια ευρώ των πληρωμών στο κεφάλαιο 4. Και ειδικότερα τώρα για την ανθρωπιστική βοήθεια. Ο διαθέσιμος για την ανθρωπιστική βοήθεια προϋπολογισμός κατά το 2013 αυξήθηκε κατά 410 εκατομμύρια και για τις θεσμές χρόνων και για τις πληρωμές με τον διορθωτικό προϋπολογισμό και την ε, αναδιανομή στο ιστορικό του κεφαλαίου 4 και την κινητοποίηση του μηχανισμού κατεπίγουσας βοήθειας. Για το 2014 η κατάσταση για τις πληρωμές όπως το γνωρίζουμε ήδη είναι πολύ τεταμένη όπως ήδη είπαμε. Οι μη εξοφληθήσεις αποδείξεις, οι μη λογαριασμοί μόνο για τη συνοχή και δεν αναφέρομαι σε άλλα κεφάλαια του προϋπολογισμού Θα δούμε όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία κλείσιμο των λογαριασμών, ειδικά για τη συνοχή, επαναλαμβάνω και μόνο για τη συνοχή, μένουν ανεξόφλητα 23,4 δισεκατομμύρια. Σημαντική αύξηση ανεξόπλητων ποσών σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Μίλησα για τεταμένη κατάσταση. Δεν είναι αυτό αξιοπεριέργο, ήταν, ήταν ήδη γνωστό και κατά την έγκριση του προπολογισμού. Το είχαν επισημάνει και το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή με μια κοινή δήλωση ειδικά για τις πληρωμές. Δεν θα επαναλάβω το κείμενο της ανακοίνωσης, της δήλωσης αυτής, αλλά ήταν σαφές, ήταν γνωστό. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν μια σειρά προγραμμάτων εξωτερικής βοήθειας θα αντιμετωπίσουν προβλήματα στις πληρωμές κατά τη διάρκεια του 2014 και σχετικά νωρίς μέσα στο έτος, ιδιαίτερα δε η ανθρωπιστική βοήθεια. Από πλευράς τη Επιτροπής και κυρίως της Γενικής μας Διεύθυνσης, εμείς παρακολουθούμε με πολύ μεγάλη προσοχή την κατάσταση και έχουμε προβεί μια σειρά επιλογών για κάποιες δράσεις σε συνεργασία καταρχάς με τους ε, συναδέλφους από τις αρμόδιες γενικές διευθύνσεις λαμβάνουμε, ή με την αρμόδια γενική διεύθυνση λαμβάνουμε μέτρα ώστε να ε, διαχειριζόμαστε το επίπεδο των συμβάσεων και να το αναπτύσσουμε στη διάρκεια του έτους κατά τρόπον ώστε να αξιοποιούνται όσο το δυνατόν καλύτερα τα διαθέσιμα ποσά, τα οι διαθέσιμες προβλέψεις από τις δεσμεύσεις υποχρεώσεων, ειδικά για την ανθρωπιστική βοήθεια. Η επιλογή ήταν να προχωρήσουμε σε δύο στάδια για τη διάρκεια του έτους, μειώνοντας και τα επίπεδα προχρηματοδότησης όπως αυτά έχουν ε, διανεμηθεί στις διεθνείς ε, οργανώσεις. Και για να αντιμετωπίσουμε τα συγκεκριμένα προβλήματα στις πληρωμές, θα χρειαστεί να αξιοποιήσουμε μια σειρά από μέσα, σε τεχνικό επίπεδο. Πρώτον, θα θεσπίσουμε, ήδη έχουμε ξεκινήσει να θεσπίζουμε και θα δείτε το σχετικό αίτημα για, το, για τη μεταφορά των κονδυλίων. Θα αρχίσουμε λοιπόν να χρησιμοποιούμε το μέσο των εμβασμάτων που επιτρέπουν σε αυτό το στάδιο χρονικά να έχουμε στη θέσή μας τα απαραίτητα για την ανθρωπιστική βοήθεια ποσά και αργότερα με στη διάρκεια του έτους με έναν διορθωτικό προπολογισμό θα επιστρέψουμε τα ποσά, θα, θα αποζημιώσουμε αυτούς που μας τα έχουν ε, διαθέσει. Γιατί όπως είπα, οι περιορισμοί αυτή, η στενότητα αυτή αφορά όλες τις θέσεις και κυρίως την ανθρωπιστική βοήθεια. Και έτσι έχουμε δύο αιτήματα για εμβάσματα για 150 εκατομμύρια ευρώ σε επιστώσεις πληρωμών, ανθρωπιστική βοήθεια, τον ΤΕΚ 6 και για το μέσον για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον ΤΕΚ 10. Άρα πρόκειται για μέτρα που θα εκφραστούν σε εμβάσματα. Εφόσον δεν χρειαστεί, θα αξιοποιήσουμε και το μέσο της κατεπίγουσας βοήθειας, εάν δεν υπάρξουν στη διαθέσή μας βραχυπρόθεσμα άλλα μέσα. Αργότερα δε μέσα στο έτος θα αξιοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα μέσα τη συνολική μεταφορά των κονδυλίων, την αναδίπλωση, αναδιανομή των ε, κονδυλίων στο βαθμό που έχουμε τη δυνατότητα για πληρωμές όπου είναι δυνατόν και σε σχέση με την ε, υλοποίηση του προπολογισμού η προώθησή μας από πλευράς της Επιτροπής είναι να απευθύνουμε έτοιμα για κινητοποίηση του περιθωρίου που είναι ακόμα διαθέσιμος προς ε, το νοτοτόριο των πληρωμών. Ξέρετε ότι έχουμε ένα περιθώριο 711 εκατομμυρίων, τουλάχιστον όσο προκύπτει από την κοινή ανάγνωση των ε, λογαριασμών των υπολογισμών από πλευράς Επιτροπής και Κοινοβουλίου. Και θα προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατό μηχανισμό ευελιξίας από το πολιτισμικό οικονομικό πλαίσιο, από την ε, διοργανική συμφωνία, οτιδήποτε δυνατότητα υπάρχει θα αξιοποιηθεί. Ιδίω δε, εφόσον χρειαστεί, θα αξιοποιηθεί και η δυνατότητα του περιθωρίου για κατές περιπτώσεις που προβλέπει το άρθρο 13 του κανονισμού για το δημοσιονομικό πλαίσιο, το πολιτές πλαίσιο. Αυτά. Εντάχει υπενθύμηση του ιστορικού τη τρέχουσα κατάσταση και των προοπτικών ω προ την κινητοποίηση μια σειρά μέσων, η οποία θα αναπτυχθεί μέσα σε ένα χρονοδιάγραμμα από σήμερα μέχρι και τουλάχιστον από πλευρά τη Επιτροπή οι πρωτοβουλίε μα θα αναπτυχθούν μέχρι το καλοκαίρι, πριν το καλοκαίρι δηλαδή, ελπίζοντα ότι η Δημοσιονομική Αρχή, Συμβούλιο και Κοινοβούλιο θα μπορέσει να ανταποκριθεί κατά τρόπο αποτελεσματικό και ταχύ στις, στα αιτήματα που θα καταθέσει η Επιτροπή. Και σε αυτό δεν αμφιβάλλουμε καθόλου για την υποστήριξη που θα μα προσφέρει το Κοινοβούλιο. Εάν επιτρέπετε όμω, ο συνάδελφο κ. Σέρενσεν θα μπορούσε να συνεχίσει μετά από μένα. Ευχαριστώ. Όντως, για να συνεχίσω από εκεί που καταλήξατε, έχετε αντιληφθεί πλήρω ότι η Επιτροπή Προϋπολογισμών ασχολείται με το πρόγραμμα, αυτό το πρόβλημα και με την ομάδα παρακολούθηση αλλά και προηγουμένως με ακρόαση δύο επιτρόπων είναι διότι ανησυχούμε ε, σφόδρα για τις ε, πιστώσεις πληρωμών που Υπάρχει πρόβλημα παντού σε όλες τις θέσεις του προπολογισμού, αλλά διαφέρουν και επιπτώσεις. Καμιά φορά μπορεί να είναι δραματικές, ε, ανάλογα με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επίσης, επειδή λύγει και η θητεία του Κοινοβουλίου και θα ανανεωθεί το Κοινοβούλιο, μετά τις ευρωεκλογές, επί σειρά εβδομάδων θα είναι κάπως παραγκονισμένο το κοινοβούλιο και υπάρχουν κατεπίγουσες πολιτικές όμως που δεν μπορούν να περιμένουν. Εμείς θέλουμε να είμαστε βέβαιοι ότι θα είναι εξασφαλισμένες όλες οι διαθέσιμες ε, διαδικασίες και θα εκτελούνται έτσι ώστε να περιορίζεται όσο γίνεται, για να μην πω να ε, καλυφθεί πλήρως ε, αυτό το κενό και οι ανετικές συνέπειες να αποσοφηθούν. Είναι αναπόφευκτη αυτή η δημοκρατική παρένθεση των εκλογών τέλη του διαστήματος αυτού της Άνοιξης. Ο Γενικός ε, Διευθυντής του Γραφείου Ανθρωπιστικής Βοήθειας νομίζω θα μπορέσει να συμπληρώσει με τις δικές του πληροφορίες. Ευχαριστούμε κύριε Γενικέ. Ε, κύριε Σάνουσεν, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, ε, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη γιατί έφερα διαφάνειες αλλά διαπιστώνω ότι πρέπει να έχετε τρομερή όραση για να μπορέσετε να παρακολουθείτε. Μα έχω, αλίμονο. Ε, έχω, έχω, καλά μάτια. Μπορείτε να παρακολουθήσετε. Ούτε εγώ δεν μπορώ να τα δω αυτά, αλλά εγώ είμαι προνομίχος, διότι τα έχω μπροστά μου σε κείμενο. Ε, πάση περιπτώσει, επί της ουσίας, νομίζω ότι ε, μπορώ να σας παρουσιάσω μία επισκόπηση του θέματος αρκετά ε, συνοπτικά. Καταρχάς, συμφωνώ με τη συνάδελφό σας, την κυρία Αν ότι πραγματικά είμαστε σαν μια χιονοστιβάδα, ε, χρόνο με το χρόνο ε, συσσωρεύεται το υπόλοιπο προς εκαθάριση και η καθυστέρηση στις πληρωμές. Τι σημαίνει αυτό. Υπάρχουν ανεξόφλητοι λογαριασμοί, οι οποίοι όμως είναι οφειλόμενοι. Ε, βλέπετε πως έχει κατάσταση εδώ στη γραφική παράσταση και έχουμε φτάσει πια σε ένα τέτοιο σημείο που χωρίς ενίσχυση και σας ευχαριστώ πάρα πολύ πολύ ευγνώμων προς τον κύριο Ζωνζόν και τους συναδέλφους ε, της Γενικής Διεύθυνσης Προϋπολογισμού αλλά και των υπολείπων γενικών διευθύνσεων όπου εργάζονται οι συνάδελφοι. Χωρίς αυτή την ενίσχυση το προσεκαθάριση υπόλοιπο θα ήταν πολύ υψηλότερο από την ανάληψη υποχρεώσεων σε αιτήσια βάση του προπολογισμού για να μην πω και για τις πιστώσεις πληρωμών που θα ήταν πολύ μεγαλύτερη διαφορά. Αυτό δεν πειράζει καταρχήν να είναι μεγάλος ο κύκλος του προγράμματος, αλλά εμείς τώρα θα πρέπει να εκαθαρίσουμε και να εξοφλήσουμε μέσα σε 18, 12-18 το πολύ 24 μήνες. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε τρόπος παράτασης ή αναβολής, διότι εκείνοι που διαχειρίζονται σε καθημερινή βάση τα προγράμματα χρειάζονται τα χρήματα ε, διαφορετικώς θα πτωχεύσουν. Αυτό δεν ισχύει ακριβώς για τους οργανισμούς των ΗΕ, αλλά υπάρχουν και οργανισμοί των ΗΕ με τους οποίους έχουμε ε, συμβάσεις και έχουμε και συμβατική υποχρέωση να τους προκαταβάλουμε 80% για το Παγκόσμιο Επιστημιστικό Πρόγραμμα, για την ύπατη αρμοστία, για τους πρόσφυγες κτλ. Και εγώ θα πρέπει γονεί γονίπετής κάθε φορά να τους παρακαλώ ε, να μας δώσουν μια διορία και το κάνουν γιατί είναι πολύ γενναιόδοροι, αλλά υπάρχουν και όρια. Ε, στη γενεοδορία και στη δική μου οικεσία, γιατί ουσιαστικά συσσωρεύεται έτσι χρέος για την επόμενη περίοδο και αυτό είναι το πραγματικό μου δίλημα. Διότι έχουμε ένα σωρευτικό εδώ αποτέλεσμα. Βλέπετε τη διαφορά ανάμεσα στις δύο πράσινες στήλε στην γραφική παράσταση, που είναι η διαφορά ανάμεσα στην ανάληψη χρεώσουν και στις πληρωμές που χρόνο με το χρόνο μετακυλείεται αυτό και θα πρόσθετα και εδώ ότι υπάρχει και η ετήσια ενίσχυση που ε, καταβάλλεται και πολύ συχνά μας δίδεται και ευχαριστώ και πάλι ε, τους καλούς συναδέλφους και χάρη σε αυτούς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, παίρνω κονδύλια για την υπόθεση ας πούμε της Συρίας φέτος αλλά αυτό είναι που χρεώσεων, δεν ακολουθούν οι πληρωμές. Και αυτό είναι λοιπόν τώρα ένας βραχνάς που έχουμε να μεταφέρουμε στο επόμενο διάστημα και ένα βάρος για να είμαι ειλικρινής μέχρι πέρυσι κάπως θα καταφέρναμε να τα βγάζουμε πέρα διότι κανονικά στα τέλη του έτους ε, υπάρχουν κάποιες πιστώσεις πληρωμών που ε, κυκλοφορούν, περισσεύουν, γίνονται μεταφορές πιστώσεων και τα βγάζουμε πέρα. Αλλά πέρυσι αυτή η πηγή χρηματοδότησης ε, απλούστατα στέρεψε και ήταν πάρα πολύ δύσκολο ακόμα και με τη μεγάλη βοήθεια της Γενικής Διεύθυνσης Προϋπολογισμού να κάνουμε αρκετές μεταφορές πιστώσεων και να κινητοποιήσουμε τα κονδύλια που χρειαζόμαστε για να καλυφθεί το έλλειμμα το οποίο είχαμε συσσωρεύσει. Πρέπει να σας πω, για να είμαι και δίκαιος και ειλικρινής, ότι πραγματικά μας υποστήριξαν πάρα πολύ, όντως και σας ευγνωμονώ και σας ιδιαιτέρως, αλλά το πρόβλημα έχει αυξηθεί τώρα σε τέτοιο βαθμό που όσο σημαντική και ενίσχυση και γενναία δεν ήταν επαρκής. Ε, και εσείς οι ίδιοι ε, το εντοπίσατε αυτό το πρόβλημα, διότι προτείνατε ε, πολύ σοφά πέρυσι έξτρα ενίσχυση στις πιστώσεις πληρωμών για το 2014, τον προϋπολογισμό του. Και επίσης προτείνατε να προσθεθούν περισσότερες πιστώσεις πληρωμών στο αποθεματικό για την ε, κατεπίγουσα βοήθεια. Δηλαδή περισσότερες πληρωμές από ό,τι αναλήψεις ε, υποχρεώσεων. Πολύ δημιουργικό αυτό και εμπνευσμένο. Δυστυχώς ε, να βάγισαν οι τροπολογίες αυτές. Εάν είχαν περάσει, θα ήταν πολύ πιο άνετη η δική μου δουλειά στο μικρό μου επίπεδο και ίσως θα μπορούσαμε να τα είχαμε βγάλει πέρα με έναν τρόπο πιο παραγωγικό. Πέρυσι που καταλήξαμε. Ακριβώς επειδή έπρεπε να ζητήσουμε από ΜΚΟ να αναβάλουν τις πληρωμές, δεν τους προκαταβάλαμε το 80%, τους είπαμε θα πάρετε 40% για αρχή και μετά ελπίζουμε όταν θα ρεύσουν τα χρήματα μετά τον Νοέμβριο, με το καλό θα πάρετε και τα υπόλοιπα. Πλην όμως ε, κάποια από τα χρήματα αυτά ήρθαν μόνο με το φετινό προπολογισμό και θα καταλάβετε ότι όταν εγώ πρέπει να προκαταβάλω τον Ιανουάριο ε, σε μετρητό, ήδη μου αφαιρούν τα χρήματα που θα ήθελα εγώ να δαπανίσω για νέες συμβάσεις στο νέο χρόνο. Δεν υπάρχει τρόπος αυτό να αποφευθεί, απλώς να το αναγνωρίσουμε ως γεγονός. Αυτές οι ελλείψεις και τα ελλείμματα πληρωμών θα πρέπει να αντιμετωπιστούμε κάποιο τρόπο. Και ε, είπε προηγουμένως ο Γενικός Διευθυντής ότι ε, προσβλέπουμε στην καλή θέληση της δημοσιονομικής αρχής ότι θα ακολουθήσουν ροές κεφαλαίων, αλλά μέχρι τότε θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα στερέψουν τα χρήματα μέχρι να εγγραφούν νέα στον προϋπολογισμό. Έτσι έχει η κατάσταση. Επίσης ε, βλέπετε αυτή τη γραφική παράσταση με τα διάφορα ε, κομμάτια της τούρτα στο κίτρινο και το γαλάζιο είναι το σύνολο των πιστώσεων πληρωμών που έχουμε στη διάθεσή μας. Και τι μας κάνει εντύπωση εδώ. Ε, τι νέο που για μένα δεν είναι είδηση γιατί το έχω αντιληφθεί εδώ και καιρό είναι ότι όλα τα χρήματα που είναι στη γαλάζια φέτα καλύπτουν τις υποχρεώσεις μας για το 2013 και το 2012. Δηλαδή, πριν αρχίσουμε καν να συνάπτουμε νέες συμβάσεις και τα λοιπά, θα πρέπει να εξοφλήσουμε κατά τη διάρκεια του έτους, καθόλου το 14, όχι τον Ιανουάριο, καθόλου τη διάρκεια του έτους, και αυτό είναι προβλέψιμο ως δαπάνη. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να αρχίσω να δαπανώ αυτά τα χρήματα, διότι θα ήταν εκ μέρους μου ε, ανεύθυνη η οικονομική διαχείριση. Ε, η κίτρινη φέτα είναι επίσης και περισσότερο περιοριστική θα έλεγα, διότι είναι η καθυστέρηση στις ανεξόφλητες ε, οφειλές που έχουμε την 1η Ιανουαρίου και πρέπει να σας πω ότι αυτό το εξοφλήσαμε μόλις μπήκε στο κονδύλι το ποσόν ε, στον προπολογισμό του 2014. Και μετά έχουμε βάλει στην άκρη ένα ποσό για τα πάγια έξοδα ε, που είναι οι δαπάνες για το προσωπικό επιτόπου ε, για ε, το ΕΚΟ. Γιατί θέλουμε να καταστρέψουμε και την υποδομή επιτόπου επειδή έχουμε κάποια ταμιακή δυσκολία. Υπάρχουν κάποια πάγια ή παγωμένα κονδύλια που θα πρέπει να τα... Είναι ασυμπίεστες δαπάνες ας πούμε. Είναι λιγότερο από 100 εκατομμύρια ευρώ στην αρχή του έτους. Θα έπρεπε να τα βάλω στην άκρη αν έχω ένα έτσι, ειλικρινή προπολογισμό. Βεβαίως η ρευστότητα πλέον είναι μεγαλύτερη διότι δεν χρειάζεται να δαπανηθούν στις αρχές του έτους όλα αυτά τα χρήματα όπως και δεν τα δαπάνησα. Έχουμε ακόμα ε, μετρητά αλλά αν θέλουμε να φτάσουμε κοντά ε, περίπου στις υποχρεώσεις που έχουμε για εφαρμογή ε, χρειάζομαι ε, κάποια ενίσχυση της ρευστότητας. Και έρχομαι στην επόμενη διαφάνεια που σίγουρα δεν βλέπετε και λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά για να μην μακρηγορώ, ήδη σήμερα Νομίζω είμαστε σε θέση να δώσουμε ευχάριστα νέα, διότι χάρη στους συναδέλφους μου, στη Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ, στη Γενική Διεύθυνση Ρέγγιο και στη Γενική Διεύθυνση Διεύρυνσης καταφέραμε με κάποιο τρόπο να βρούμε κάποιες προκαταβολές που μου δίνουν για ε, τις πιστώσεις πληρωμών γιατί ξέρουν ότι δεν έχουν τόσες ε, άμεσες και οξύες ανάγκες όπως εγώ και μάλλον έχετε λάβει, θα έπρεπε να έχετε λάβει μια ε, πρόταση μεταφορά πιστώσεων 150 εκατομμυρίων που για μένα είναι ζωτική σημασία, διότι αυτό θα μου επιτρέψει να συνεχίσω τις συμβάσεις μου με τον τρόπο και την ταχύτητα που κάνουμε αυτό το καιρό. Λοιπόν, για να καλύψουμε όλες τις ανάγκες χρηματοδότησης και να τιμήσουμε ας πούμε τις υποχρεώσεις μας σε ένα εύλογο διάστημα και λέω εύλογο γιατί δεν είναι η τέλεια λύση αλλά τουλάχιστον για να επιβιώσουμε όπως και πέρσι περίπου τα βγάλαμε πέρα θα σας ήμουν ιδιαίτερος ευγνώμων εάν εκτός από τα 150 μας δίνατε άλλα 250 ε, κάποια μορφή ε, διορθωτικού προπολογισμού. Και ο κύριο Ζανζόν, ο κύριος Γενικός, ε, είπε ότι ε, το έχουμε υπόψη μας, δεν χρειάζεται να μπούμε τώρα σε λεπτομέρειες, αλλά αυτό θα σας παρακαλούσα να ε, σκεφτείτε, γιατί σε αυτό προσβλέπω. Και προφανώς, ε, τη στιγμή που θα κάνει την πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλα θα έχουν ξεκαθαριστεί στο δικό μας θεσμικό όργανο, νομίζω θα είμαι σε μια αρκετά βολική θέση να αρχίσω να υπογράφω συμβάσει για την περίφημη δεύτερη φάση. Αλλά θα πρέπει όλα αυτά να είναι αρκετά έτσι, γερά και στιβαρά. Δεν θέλω να βρεθώ σε μια κατάσταση που για κάποιου μυστήριους λόγους να έχουμε υπογράψει συμβάσει, ιδιαίτερα με μη κυβερνητικέ οργανώσει που εξαρτώνται από εμάς και μετά να είναι το ταμείον μείον. Καταλαβαίνετε ποια θα είναι η θέση μας θα είναι χειρότερα από το να σταματήσω να υπογράφω και να προκαταβάλω. Λοιπόν, αυτά τα 150 εκατομμύρια πιστώσεις, μεταφορά πιστώσεων και τα 250 θα με βοηθήσουν να τα βγάλω πέρα για φέτος. Ξέρετε, όπως και εσείς είστε έτσι πολύ υπεύθυνοι διαχειριστές οικονομικοί, και αυτό θα, στο τέλος του χρόνου θα με φέρει ένα υπόλοιπο όπως είχα και πέρσι, δηλαδή περίπου 160 εκατομμύρια ευρώ. Φέτος κατάφερα να ε, επιβιώσω ας πούμε και ε, του χρόνου επίσης αλλά δεν θα ε, συνιστούσα σε κανένα να αυξηθεί γιατί απλώς αυτή η χιονοστιβάδα συνεχίζει την πορεία της και αυξάνει το μέγεθός της και δεν θεωρείται αυτή η διαχείριση υπεύθυνη. Συμπέρασμα, θα πρέπει να συνεργαστούμε με τη δική σας Επιτροπή και με την επόμενη Επιτροπή Προϋπολογισμών μετά τις ευρωεκλογέ. Εμείς είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε, αλλά καταλαβαίνετε ότι ανακύπτουν κάποια ερωτηματικά. Πώς φτάσαμε εδώ και τι μπορεί να γίνει στο μέλλον και τι πρέπει να γίνει για να αποφύγουμε παρόμοιες καταστάσεις και προβλήματα. Έχουμε κάποιες προτάσεις εδώ, βέβαια δεν είναι θαύματα, είναι λογική αυτά που προτείνουμε. Θα πρέπει να αναρωτηθούμε εάν είναι υγιής αυτή η κατάσταση, να συνεχίσουμε να δημιουργούμε ένα υπολογισμό για ανθρωπιστική βοήθεια, όπου η ανάληψη υποχρεώσεων είναι πάντα πολύ μεγαλύτερη από τις πληρωμές. Ή υπολείπονται ε, συνεχώς οι πληρωμές. Στο παρελθόν κάτι τέτοιο λειτουργήσε, γιατί κάπως στα τέλη του έτους συμμαζεύαμε λίγο ε, κάποιες πιστώσεις ε, από αλλού που περίσευαν, αλλά εάν επαναληφθεί αυτό επειδή και οι πόροι φθήνουν και σπανίζουν όλο και περισσότερο θα έχουμε ε, προβλήματα στο μέλλον να συνεχίσουμε αυτή την τακτική. Και χαίρομαι πάρα πολύ που η ιδέα αυτή υιοθετήθηκε και ε, στο ψήφισμα για την απαλλαγή. Είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να εργαστούμε σε αυτή τη βάση. Μία άλλη ιδέα που κυκλοφορεί είναι να υπάρξει ένα συγκεκριμένο ποσό που να απευθύνεται σε ανθρωπιστική βοήθεια. Τα κράτη-μέλη ενδιαφέρονται άρα για να βγάλουν χρήματα από τον κρατικό τους προπολογισμό και να τα ε, αφιερώσουν ειδικά στην ανθρωπιστική βοήθεια. Έχουμε μια πολύ καλή ε, περίπτωση η γαλλική κυβέρνηση, περίπου 20 δισεκατομμύρια έχει ε, απελευθερώσει για συνεργασία μαζί μας στην ακτή Ελεφαντοστού. εκατομμύρια, συγγνώμη. Ε, αυτό είναι κάτι ίσως του απότερου μέλλοντος, αλλά ε, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και αυτή τη δυνατότητα. Θα πρέπει όμως ειλικρινά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο να συνεννοηθούν για το πώς θα έχουμε αυτές τις πιστώσεις ε, εκτός των ορίων και για τις αναλήψεις υποχρεώσεων και για τις πληρωμές. Είναι σημαντικό αυτό. Δεν μπορεί επειδή έχουμε ένα πλαφόν ξαφνικά να μην μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις επίγουσες τύπου IT κτλ. Συγγνώμη που μακρηγόρησα λίγο. Θα μπορούσα να μπω σε πολύ περισσότερες λεπτομέρειες για τη διαχείρισή μας. Έχουμε λεπτομερέστατη και σχολαστικότατη ε, αποτίμηση κάθε χώρας και κάθε σύμβασης για να δούμε ποιο είναι το πιο επίγον που ε, κινδυνεύουν ζωές, που υπάρχουν άλλοι δωρητές που μπορούν να αναλάβουν αντί για μας, για να είμαστε και σε θέση να διαχειριζόμαστε πάντα όλα αυτά τα θέματα και αυτό το σφιχτό δημοσιονομικό πλαίσιο που έχουμε. Και θα ήθελα να αποτίσω και ένα φόρο τιμή στους υπαλλήλους μου. Εκτός από τη συνήθεια τους δουλειά, έχουν αναλάβει και αυτά και είναι βαριά δουλειά. Και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ και την κοινότητα των μη κυβερνητικών οργανώσεων, γιατί και για εκείνους ήταν αντίστοιχα οδυνηρά τα πράγματα και ε, περίπλοκα. Παραμένουμε σε στενή επαφή, τίποτα δεν είναι τέλειο εδώ, αλλά θέλω να αποτίσω φόρο τιμής και στην κατανόηση αλλά και στην υπομονή τους. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστώ <clears throat> τον Γενικό Διευθυντή. Θα ήθελα να σας θέσω ένα ερώτημα. Μπορείτε να μας δείξετε παρακαλώ την σελίδα 4, τον πίνακα της σελίδας 4. Θέλω να είμαι βέβαιος ότι κατάλαβα σωστά πράγματι θα πρέπει να τα βλέπει κανείς αυτά πιο προσεκτικά. Λοιπόν, για τις ανάγκες για Μέσα το 2014. Αυτές είναι οι ανάγκες. Στη μέση είναι οι διαθέσιμες πληρωμές για το 2014, χάρη στις πρώτες προσπάθειες μεταφοράς. Όχι, πριν τις μεταφορές. Λοιπόν, υπάρχει μια τεράστια διαφορά εδώ και έλλειψη πιστώσεων. Και οι δημοσιονομικές επιλογές. Το πράσινο 776 είναι ακριβώς η πρίκα σας από τον προϋπολογισμό του 14, η αρχική. Εσείς θα θέλατε να προσθεθούν εκεί 150 εκατομμύρια μεταφορές, το λεγόμενο TEC 6, Ελπίζεται παράλληλα έναν διορθωτικό προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια, αυτό το ανέφερε και ο Γενικός Διευθυντής, κάτι το οποίο θα σας επιτρέψει να κλείσετε το χρόνο με μια καθυστέρηση πληρωμών αντίστοιχη του προηγούμενου έτους, κάτι το οποίο είναι βιώσιμο και δεν είναι σκανδαλώδες και τεράστιο είναι διαχειρίσιμο λέει ο Γενικός Διευθυντής αλλά η κατάσταση αυτή δεν πρέπει να συνεχιστεί. Αλλά θα τα βολέψουμε για φέτος. Λοιπόν το ερώτημά μου είναι το εξής. Παρουσιάσατε πάρα πολύ καλά τα κατεπήγοντα προβλήματα πληρωμών τα οποία είχατε. Μας παρουσιάσατε τις δράσεις οι οποίες γίνονται αντικείμενο διαχείρισης άμεσα από πλευρά σας ή από μικιό συνδεδεμένες με σας και κάποιες δράσεις με τις οποίες έχετε συμβατική σχέση με τα Ηνωμένα Έθνη και είπατε ότι τα Ηνωμένα Έθνη μπορείτε να διαπραγματευτείτε μαζί τους για κάποιες καθυστερήσεις από πλευράς μας, αλλά αυτό έχει κάποια όρια. Ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή, ποιες είναι οι τάξεις μεγέθους του χρέους που έχουμε, που έχετε απέναντι στα Ηνωμένα Έθνη και άλλες διεθνείς οργανώσεις. Αυτό ανταποκρίνεται στη γνωστή καθυστέρηση, μιλάμε για επιπλέον ποσό. Μια τάξη μεγέθους για να καταλάβουμε τι αντιπροσωπεύει στο σύνολο του προϋπολογισμού. Κοιτάξτε, αυτό είναι πρόχειρο εδώ που λέω, αλλά ο μισός μας προϋπολογισμός αφορά τους διεθνείς οργανισμούς, διαπραγματευθήκαμε μαζί τους και αντί να τους δώσουμε προκαταβολή το 80% το οποίο δικαιούντο, κατεβήκαν στο 40% σε επίπεδο προχρηματοδότησης. Παραμένει λοιπόν άνω του 50%. το 50% του 50% είναι ένα τέταρτο, δηλαδή είμαστε περίπου στο συνολικό ποσό των 160 εκατομμυρίων. Θέλω να ευχαριστήσω αυτούς τους διεθνείς οργανισμούς. Κάποιοι από αυτούς είπαν μη μας δώσετε καθόλου λεφτά και υπογράψτε και μας πληρώνετε του χρόνου. Αυτό είναι ενδιαφέρον βέβαια αλλά και πολύ επικίνδυνο γιατί στην ουσία σπρώχνω πάλι μπροστά μου και μεγενθύνω τη χιονόμπαλα. Και μεγενθύνεται η χιονόμπαλα και θα μας πλακώσει. Πρέπει να τους πούμε λοιπόν όχι ευχαριστούμε, δεν θέλουμε την προσφορά σας, κατεβαίνω στο 40% και προχωράμε. Για να μην υπονομεύσουμε το μέλλον. Μας βοήθησαν οι διεθνείς οργανισμοί πάρα πολύ σχετικά με τους τόκους και αυτοί έχουν δικαίωμα να παίρνουν τόκους για καθυστερήσεις. Αλλά είπαν στη συγκεκριμένη περίπτωση ότι δεν θα το κάνουν. Εκεί που πληρώνουμε είναι για τις ΜΚΟ και αυτό είναι φυσιολογικό. Καταλαβαίνω λέει ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ, η μαρτυρία σας ή το επακριβεστάτη. Ε, θα δώσω το λόγο στον κύριο Μπαγκούρ. ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Γενική Διεύθυνση Συνεργασίας και Ανάπτυξης με Διευθυντής των πόρων για το 2013. Ήταν μια πολύ καλή χρονιά ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Είχαμε ποσοστό 100% εκτέλεση, είτε μιλάμε για υποχρέωση, είτε μιλάμε για πληρωμές. Πρέπει να σημειώσουμε ότι χρόνο με το χρόνο έχουμε ε, ε, έργα τα οποία δεν υλοποιούνται και σωρεύονται με 1,9 δις ευρώ από το 2009, απόκληση μεταξύ υποχρεώσεων και πληρωμών και, 1, και αυτό το 1,9 αφορά και γεννά παράγει το, τα υπόλοιπα προς εκτέλεση, το ραλ δηλαδή για τα επόμενα χρόνια. Είχαμε ραλ στο τέλος του 2013 συνολικά 15,5 δις Αυτά λοιπόν τα υπόλοιπα. έχουν σαν αποτέλεσμα προς το τέλος ε, του 2013, όπως και για τις άλλες πολιτικές, ε, κάποια έλλειψη ποσών που μας υποχρέωσαν να αναβάλουμε για τις αρχές του 2014 την πληρωμή ε, λογαριασμών μέχρι 300 εκατομμύρια ευρώ. Για το 2014 τώρα έχουμε ένα προϋπολογισμό ο οποίος θα μας επιτρέψει να εξασφαλίσουμε τη διαχείριση και των προηγούμενων προγραμμάτων, αλλά και νέων προγραμμάτων. 11 Μαρτίου του 2014 συγκεκριμένα ε, εγκρίθηκε το σύνολο των δημοσιονομικών μέσων για την περίοδο 2014-2020 και δημοσιεύθηκαν στις 15 Μαρτίου τα σχετικά κονδύλια. Όπως είχαμε συμφωνήσει με το Κοινοβούλιο, έχουμε προχωρήσει σε στρατηγικό διάλογο με τις Επιτροπές ΔΕΒΕ και ΑΦΕΤ ο προσεχής στρατηγικός διάλογος προβλέπεται για αύριο, 1η Απριλίου και είμαστε έτοιμοι να επεξεργαστούμε και να καταθέσουμε για την Επιτροπολογία το σύνολο των πολιετών προβλέψεων πριν τις τεχνές διακοπές. Άρα πρώτο ε, πολιετές ε, σχέδιο αλλά και εγκρίσεις για ορισμένες περιπτώσεις αναμένεται να είναι έτοιμα πριν τις διακοπές ή πάντως πριν το τέλος του έτους. Για το 2014 έχουμε υποχρεώσει σε ύψος 4,7 δις και πληρωμές σε επίπεδο 3,4. Έχουμε δηλαδή 1,3 εκατομμύρια ευρώ, ε, δισεκατομμύρια ευρώ απόκληση, που σημαίνει ότι εάν δεσμεύσουμε τα ποσά και πληρώσουμε ό,τι χρειάζεται, θα μας μείνει ένα υπόλοιπο ραλ 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ, εάν όλα πάνω όπως προβλέπονται. Η δική μας διαπίστωση είναι ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα ως προς τις πιστώσεις υποχρεώσεων του 2014, όπως ανέφεραν άλλωστε, ανέφερε άλλωστε και ο Γενικός Διευθυντής ΕΚΟ και ο Γενικός Διευθυντής ε, του Προϋπολογισμού, έχουμε αναπτύξει την ιστορική αλληλεγγύη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής και έτσι έχουμε προκαταλάβει για την ανθρωπιστική βοήθεια, για το κεφάλαιο 4, τα πόσα για τις πληρωμές. Έχουμε ωστόσο εμείς δικά μας προβλήματα προ τι πιστώσει πληρωμών και προχωρούμε με πολύ προσεκτική διαχείριση, η οποία σημαίνει καταρχά ότι δίνουμε τα εμβάσματα γραμμή με τη γραμμή, ε, κώδικα με τον κώδικα στον προπολογισμό, ώστε να μην βρεθεί καμία γραμμή χωρίς κονδύλια. Έχουμε ένα ποσοστό εκτέλεσης πληρωμών σε ύψος 65% για τα ανθρώπινα δικαιώματα σήμερα, για την αναπτυξιακή βοήθεια 67%, για την υποστήριξη κοινωνίας των πολιτών 50%, με σημερινά στοιχεία. Δηλαδή αξιοποιούμε πιστώσεις πληρωμών για κάποια κονδύλια τα οποία τον Νοέμβρη το Δεκέμβριο ολοκληρώνονται για να ενισχύσουμε ε, ανθρώπινα δικαιώματα, ανάπτυξη ή υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών. Ιδιαίτερα δε ορίζουμε και προτεραιότητες ανάλογα με τις πληρωμές, προσπαθούμε δηλαδή να καταβάλουμε αυτά τα οποία αξιολογούμε ως πιο σημαντικά κονδύλια. Εάν όμως δεν δούμε βελτίωση στον προπολογισμό μέχρι του έτους, θα χρειαστεί να προβούμε σε συγκεκριμένα μέσα μέτρα, να περιορίσουμε δηλαδή την προχρηματοδότηση ακόμη περισσότερο, να καθυστερήσουμε ορισμένες αναλήψεις συμβατικών υποχρεώσεων και ενδεχομένως να αναβάλουμε για το 2015 κάποιες πληρωμές. Πράγμα το οποίο απλώς μεταθέτει το πρόβλημα στο επόμενο έτος. Άρα και εδώ. Από τη δική μας τη διεύθυνση, τη Γενική τη αναπτυξιακή συνεργασία. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε έναν διορθωτικό προπολογισμό που θα επιτρέπει ε, να εξασφαλιστούν πρόσθετα κονδύλια μέχρι το τέλο του έτου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριο Λαμασούρ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ρωτήσω εάν στο δικό σας τομέα μακροπρόθεσμα υπάρχει μια ιδέα, μια εικόνα για μια γενική εκτίμηση των ε, ποσών που θα χρειαστούν για να εκτελεστούν οι υποχρεώσεις σχέση με τις πληρωμές γιατί τώρα έχουμε ας πούμε την ιδέα ότι αν προβλέψουμε τόσες ε, υποχρεώσεις ε, μπορούμε να έχουμε ένα 70-75% ε, σε πληρωμές και άρα προχωρούμε από τον ένα τομέα. Για την ανάπτυξη λοιπόν, αναπτυξιακή συνεργασία, έχετε κάποια αντίληψη τέτοια ή μια εικόνα τέτοια σε σχέση με αποφάσεις που έχει λάβει και το Κοινοβούλιο. Βέβαια για την περίοδο 2014-2020 έχουμε μείνει ε, στα όρια αυτής της, της ε, επιλογής του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Δεν εκτελούμε βεβαίως κατά 100% όλες τις αποφάσεις για χρηματοδότηση που έχουν ληφθεί για διάφορους λόγους. Μερικές φορές χρειάζεται να κάνουμε διαφορετικές επιλογές ανάλογα με τις υποδομές, με την κατάσταση των υποδομών ή αλλαγή πολιτικής ενδεχομένως στα κράτη εταίρους που μας αναγκάζουν να αναθεωρήσουμε τον προγραμματισμό και ενδεχομένως να καταργήσουμε κάποια ή να ματαιώσουμε κάποια προγράμματα ή όταν διαπιστώνουμε ότι κάποια προγράμματα δεν αποφέρουν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και έτσι τα ε, σταματούμε. Μια εκτίμηση λοιπόν, αρκετά αδρή θα έλεγα, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι χρειαζόμαστε 85 με 90% περίπου των σε ε, πιστώσεις πληρωμών σε σχέση με τις υποχρεώσεις. Καλώς λέω πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Και τελευταίος ο μελετής εκ μέρους Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Μάργκε. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Είμαι υπεύθυνο της υπηρεσίας που ασχολείται με τη μέσα για την εξωτερική πολιτική. Ιδιαίτερα ασχολούμεθα με το μέσο το σχετικό με τη σταθερότητα και την ειρήνη ε, μια προσπάθεια της Ένωσης να ανταποκρίνεται σε σειράξεις στον κόσμο. Το μέσο αυτό έχει σαν στόχο την άμεση δράση και αποτελούμε συνήθως την πρώτη παρέμβαση της Ένωσης ε, υπέρ των πληθυσμών που έχουν χτυπηθεί από σειράξεις πριν τεθούν σε λειτουργία άλλα μέσα που απαιτούν μεγαλύτερη περίοδο προετοιμασίας. Ε, είναι μικρής διάρκειας οι παρεμβάσεις μας, 18 μήνες κατά μέσο όρο και οι εταίροι μας έχουν ανάγκη από άμεση ταμιακή διευκόλυνση. Ήδη από τη συνθήκη της Λισαβόνας προσπαθούμε να ενισχύσουμε την παρουσία σας μας στον κόσμο και έχετε και ένα κατάλογο των δράσεων για το Μάρτιο, Ουκρανία, Συρία, Ιράν, Σουδάν, Νότιο Σουδάν και Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Σχετικά με τις ελλείψεις πιστώσεων πληρωμών, στην παρούσα φάση έχουμε καταναλώσει ήδη το 70%, επαναλαμβάνω το 70%, 102 εκατομμύρια. Όταν ξεκινήσαμε είχαμε καθυστερήσεις ε, για το 2013 βέβαια, για να διασφαλίσουμε τις κατεπίγουσες παρεμβάσεις τις οποίες αναφέρθηκα, θεωρούμε ότι το μέσο σταθερότητας θα έχει ανάγκη τον Ιούνιο-Ιούλιο μια ενίσχυση 50 εκατομμυρίων. Ελπίζουμε λοιπόν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα λάβει υπόψη τις ανάγκες του μέσου αυτού ε, στις επόμενες μεταφορές και είμαι στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ακούσατε όλοι τις παρεμβάσεις των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα θέλατε να κάνετε κάποιο σχόλιο ή να θέσετε κάποια ερώτηση. Η κυρία Ισηγήτρια, φυσικά πρώτη. Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους, λέει η κυρία Γένσεν, αυτό που είναι αστείο λίγο είναι ότι οι τομείς οι οποίοι φύγονται ε, κυρίως είναι σχετικά περιορισμένοι. Μιλάμε για ε, μικρά ποσά, τα οποία κάνουν εξαιρετικό καλό βέβαια, για τα αναπτυξιακά προγράμματα οι ανάγκες δεν είναι τόσο μεγάλες γιατί πρόκειται για προγράμματα τα οποία έχουν ε, την δυνατότητα να εξελιχθούν και να αναπτυχθούν με μεγαλύτερη χρονική άνεση. Για λόγους που εξηγήθηκαν ήδη. Λοιπόν αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να είμαστε, να συνειδητοποιήσουμε την κατάσταση και να επιμείνουμε λέγοντας πως ε, για τόσο μικρά ποσά είναι πραγματικά λυπηρό η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην μπορεί να τηρήσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει. Αυτό είναι το ένα. Ταυτόχρονα ζητήσαμε ορισμένες ερωτήσεις, θέσαμε ορισμένες ερωτήσεις για τις γραμμές για την Παλαιστίνη, για τη βοήθεια για την Ούνρα και τη Παλαιστινιακή Αρχή και γι' αυτό θα ήθελα να μας δώσετε ίσως κάποιες περισσότερες πληροφορίες για την Παλαιστινιακή Αρχή. Έχουμε αρκετές εξηγήσεις στις γραπτές σας παρεμβάσεις σχετικά με την αναμενόμενη εφαρμογή, το ποσοστό απορρόφησης. Αλλά θα ήθελα να μας το παρουσιάσετε γενικά εδώ, γιατί έχουμε ένα νέο μέσο, ένα θέμα, το θέμα της Συρίας και του Λιβάνου, με τεράστιες ανάγκες ως εκ τούτου θα ήταν χρήσιμο να ακούσουμε την δική σας αξιολόγηση για το ποια είναι πράγματι η κατάσταση και τι μπορούμε να έχουμε ε, μπροστά μας διαθέσιμα και σε υποχρεώσεις και σε πληρωμές για να αντεπεξέλθουμε. Αυτή είναι η βασική μου ερώτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Ρούμπικ. Η δική μου ερώτηση έχει να κάνει με το πόσο θα ε, επιδράσουν όλα αυτά σε μελλοντικά έργα. Είχαμε σύστηση με τον Επιτρόπο Έτιγκερ ε, το θέμα ότι στα πιο, στις πιο φτωχές περιοχές της ε, Αφρικής θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε όχι μόνο έργα όπως εγκατάσταση φωτο, φωτοκυταρικών εγκαταστάσεων αλλά και ε, τεχνογνωσία και γνώση και της χρήσης της ε, τεχνολογίας. Και είχε υποθεί επίσης ότι μπορούσαμε να έχουμε συνέργειες, ε, συνεργατικές δράσεις με το Βατικανό είτε με, τους, με τα Ηνωμένα Έθνη. Υπάρχει κάποια πρόοδο σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ποιος θέλει να απαντήσει. Ε, ευχαριστώ. Μιχαήλ Κέλλερ. Είμαι Διευθυντή αρμόδιο για θέματα γειτονία. Η κυρία Γέννησεν αναφέρθηκε στην Παλαιστίνη και τη Συρία. Πολύ φορέ λοιπόν σα δώσω κάποια στοιχεία για να απαντήσω. Όπω είπε και ο Γενικό Διευθυντή για την ανθρωπιστική βοήθεια, στον τομέα αυτό υπάρχει ανάγκη για πιστώσεις πληρωμών, γιατί περισσότερες από αυτές τις ε, δράσεις ε, υλοποιούνται από τα Ηνωμένα Έθνη και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Οι ιδιαίτεροι μη κυβερνητικές οργανώσεις δεν διαθέτουν τα μέσα εκείνα τα οικονομικά που θα τους επέτρεπαν να προχρηματοδοτήσουν τα έργα. Από το μέσον γειτονία και ιδιαίτερα για τη Συρία, η εικόνα δεν είναι διαφορετική. Από πέρσι δηλαδή έχουμε 280 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τη Συρία που δεσμεύτηκαν σε πιστώσει υποχρεώσεων για να αντιμετωπιστούν όλες οι πτυχέ της κρίσης στη Συρία με τρεις χώρες κυρίως, τον Λίβανο, την Ιορδανία και την ίδια τη Συρία ε, με βάση δε τις ανάγκες και την κατάσταση της κάθε χώρας έχουμε ε, δρομολογήσει κάθε δυνατότητα πληρωμών για να αξιοποιήσουμε να προσφέρουμε αυτή τη βοήθεια. Δηλαδή, όταν λέω κάθε δυνατότητα, για την Ιορδανία παραδείγματι, όπου υπάρχει και η δυνατότητα λόγω των γενικών κριτηρίων που έχουμε για την δημοσιονομική ενίσχυση, αξιοποιούμε τη δημοσιονομική ενίσχυση για να στηρίξουμε το Υπουργείο Εκπαίδευσης με, με 30 εκατομμύρια ευρώ για την εκπαίδευση των προσφύγων και γενικά όλων εκείνων που βρίσκονται σε ε, κοινωνίες ή κοινότητες υποδοχής λόγω της κρίσης στη Συρία. Το ίδιο και για τον Λίβανο, που η χρηματοδότηση παίρνει μέσα από τα ΕΕ και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Αυτό το αξιοποιούμε ή άλλω και για τον Λίβανο και την Ιορδανία, αλλά και την ίδια τη Συρία. Η κατάσταση λοιπόν που αντιμετωπίζουμε εμείς είναι η ίδια λίγο πολύ με αυτή που έχουν να αντιμετωπίσουν και οι συνάδελφοι της ΕΚΟ. Η μόνη διαφορά είναι ότι όταν έχουμε να κάνουμε τέτοιου είδου ε, ε, προσπάθεια, η δυνατότητες που έχουμε, όπως εδώ το Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας, έχουν πιο μακροχρόνιο προγραμματισμό οι συνάδελφοι της ΕΚΟΝ δηλαδή μπορεί να, μπορούν να τραβήξουν τις πληρωμές τους στο εξάμεινο μέχρι και ένα χρόνο ή και περισσότερο ακόμη. Ενώ τώρα εμείς για το 2013 έχουμε μπορέσει να τιμήσουμε μεν τις πληρωμές μας, ταυτόχρονα όμως βλέπουμε ξεκάθαρα ότι αυτό ήταν δυνατόν μόνο με τον προσδορισμό προτεραιοτήτων για το πού θα καταβάλουμε τις πληρωμές μας, πράγμα το οποίο σήμερα πρέπει να, να περιορίσουμε τις ε, πληρωμές μας για υποστήριξη σε άλλες χώρες το ίδιο θα απαντήσω όμως και για την Παλαιστίνη. Και αν κοιτάξετε κύριε Γένσεν με τον προπολογισμό του 2014, ότι η δημοσιονομική αρχή μας, έχει δώσει 300 εκατομμύρια ευρώ για, την, για τους Παλαιστινίους σε τρεις δόσεις, 68 εκατομμύρια για την αρχική δημοσιονομική βοήθεια, 80 για το ΟΝΡΑ, την εξειδικευμένη υπηρεσία των Εθνών για τους πρόσφυγες και 52 εκατομμύρια ευρώ για έργα που θα εκτελεστούν στα Παλαιστινιακά εδάφη. Έχουμε όμως μόνο 200 εκατομμύρια σε πιστώσεις πληρωμών, τα δύο τρίτα δηλαδή μόνο σε πιστώσεις πληρωμών σε σχέση με τις δεσμεύσεις για υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει. Έτσι λοιπόν τόσο ο πρώτος μηχανισμός ο πήγασο, όσο και οι πληρωμές στην ΟΝΡΑ θα πρέπει να καταβάλλονται σε πραγματικό χρόνο, δηλαδή παράλληλα λίγο πολύ με τον προϋπολογισμό που έχει δεσμευθεί ε, και σε επίπεδο πάρα πολύ ψηλό. Ε, μόνο μακροπρόθεσμα δηλαδή θα μπορούσαμε να καθυστερήσουμε σε ένα βαθμό κάποιες πληρωμές, αλλά για τα δύο τρίτα αυτών των πληρωμών των ε, δεσμεύσεων υποχρεώσεων καλύτερα που αφορούν τους ε, Παλαιστινίους είναι υποχρεωτικό να τα καταβάλουμε αμέσως σε πραγματικό χρόνο. Τα δύο τρίτα όπως λέω, δηλαδή τα 200 εκατομμύρια ευρώ τα οποία δεν αρκούν γιατί έχουμε και υπόλοιπο από προηγούμενα χρόνια. Και βέβαια το κύριο πρόβλημα για το οποίο κανείς δεν μιλάει είναι η Ουκρανία. Εφέτος έχετε δει τις ανακοινώσεις Επιτροπής μια εισφορά 11 δισεκατομμυρίων ευρώ που προβλέπεται, που μπορεί όμως να έχει νόημα μόνο αν καταβληθεί το ποσό ταχύτατα, όχι σε μια περίοδο 6-7 ετών, αλλά εάν ένα μεγάλο μέρος του ποσού αυτού ε, καταβληθεί ταχύτατα. Δεν είμαι σε θέση λοιπόν να σας ακριβή στοιχεία αυτή τη στιγμή, αλλά νομίζω ότι η ιδιαίτερη προσπάθεια που είναι διατεθειμένη να καταβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ουκρανία εφέτος θα ροκανίσει πολλές άλλες πληρωμές από τον μηχανισμό ε, γειτονίας. Και κάτι ακόμη, βεβαίως χρηματοδότηση ενέργειας που αποτελεί μια από τις κύριες προκλήσεις ε, που έχει να χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή. Ε, στην προκείμενη όμως περίπτωση έχουμε να χρηματοδοτήσουμε σε μεγάλο βαθμό την ε, ανάπτυξη των, της αξιοποίησης των ενεργειακών πόρων στην Αφρική από το Αναπτυξιακό Ταμείο και έτσι εκεί μπορεί το μέσον αυτό, το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο, να μας φαίνεται χρήσιμο, αλλά η κατάσταση πάλι παρουσιάζεται για προβλήματα με αυτά που σας έκανα μόλι τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ, δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ τους προσκεκλημένους μας από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα σας ζητήσω τώρα να περάσουμε στο 6, το οποίο είναι και η κατάληξη, αν θέλετε, των συμπερασμάτων της συζήτησης που προηγήθηκε για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι πληρωμές και τα υπόλοιπα προς εκαθάριση, τα ράλλα. Ε, εμείς ακούσαμε λοιπόν τα συμπεράσματα των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γι' αυτό οι συγητές μας, ο κύριος Μούλντερ και η κυρία Γένσεν, έχουν ε, προετοιμάσει ένα επεξηγηματικό σημείωμα το οποίο περιλαμβάνεται στο φάκελό σας. Ταυτόχρονα στον φάκελό σας έχετε μία επιστολή κοινή την οποία συνυπέγραψα με τον Έλμαρ Μπρόκ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων για την Ουκρανία και έχετε επίσης μια, κάποια σχέδια προφορικής ερώτησης προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Θα δώσω το λόγο στους δύο εισηγητές μας. Ο Γιάν Μιούλντα έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Άκουσα με πάρα πολύ ενδιαφέρον την προηγούμενη συζήτηση. Πάρα πολλά από αυτά τα οποία θα ήθελα να πω ε, υπόθηκαν ήδη. Αν δούμε τον προϋπολογισμό για το 2014, το Δεκέμβριο ήμασταν υπερήφανοι γιατί ήταν 6% κάτω από τα προηγούμενα χρόνια. Ήταν το καλό παράδειγμα που δείξαμε προς τα κράτη-μέλη και τα μέτρα λιτότητας. Ε, οι χώρες αυξάνουν τον προϋπολογισμό τους βέβαια, εμείς τον μειώνουμε. Στον προϋπολογισμό αυτό έχουμε περίπου ένα προβλεπόμενο περιθώριο για πρόβλεπτες ε, καταστάσεις, πέραν αυτού τίποτα. Όταν καθορίστηκε ο προϋπολογισμός και το θυμάμαι στις 2 η ώρα το πρωί στο Συμβούλιο, μας διαβεβαίωσαν οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι επαρκούσαν τα ποσά, ότι εντάξει μπορούσαμε να ήμασταν και υπερήφανοι γιατί τελικά για πρώτη φορά πήραμε περισσότερα χρήματα, ε, το Συμβούλιο έδωσε περισσότερα από όσα προβλέπεται. Θυμάμαι λοιπόν πολύ καλά ότι είχα πει τότε ότι η δική μου αίσθηση λέει ότι δεν έπρεπε να είμαστε ικανοποιημένοι, αντίθετα. Και αυτό νομίζω τεκμηριώνεται πλέον. Αν δει κανείς το πώς έχει η κατάσταση, και για να το κάνει κανείς αυτό θα πρέπει να δούμε ότι στα πλαίσια του νέου FMF έχουμε τα μέσα ευελιξίας για το τομείς όπως το Stella Field, κατεπίγουσα βοήθεια, μέσω για την παγκοσμιοποίηση. Έχουμε ένα περιθώριο 1,5 δις, το λέω λίγο βιαστικά ε, θα έλεγε κανείς ότι επαρκεί το ποσό αυτό. Αν δει όμως τον πίνακα τον οποίο σας έχω δείξει, τότε τα υπόλοιπα προς εκαθάριση ξεπερνούν τα 2 δις 21,21, 210 εκατομμύρια. Ό,τι λοιπόν ε, ε, ξεπεράσει τα ποσά αυτά φοβάμαι ότι θα δυσκολευτούμε να αντιμετωπίσουμε. Τι πρέπει να περιμένουμε λοιπόν στο μέλλον μαντεύουμε προς το παρόν σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε στο 1α, το βλέπετε στο σημείωμα το οποίο σας έχω μοιράσει, στον πρώτο τίτλο χρειαζόμαστε 1,1 δις επιπλέον. Στο 1β 36 στο 3 δεν ξέρουμε ακόμα, στο 4 οι συζητήσεις συζητάνε, ίσως χρειαστούν 400 εκατομμύρια. Θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι συνέπειες της συμφωνίας με την Ουκρανία και μαζί με τον κύριο Μπρόκ και θα πρέπει να καλύψουμε και τα της Συρίας φυσικά. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αβεβαιότητα. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε λοιπόν από εδώ και πέρα μπορούμε να ελπίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε δίκιο τον μήνα Δεκέμβριο και ότι θα κρατήσουμε μέχρι το τέλος του χρόνου. Εγώ δεν το πιστεύω. Αυτό θα δούμε τι θα γίνει. Τι επιλογές έχουμε μπροστά μας τώρα για το μέλλον. Πρώτον μπορούμε να μειώσουμε τις ε, ε, υποχρεώσεις. Δεν ξέρω αν είναι νομικά εφικτό στα πλαίσια της πολιετούς ε, δημοσιονομικής συμφωνίας δεν ξέρω αν υπάρχει μια συμφωνία και για τις υποχρεώσεις και αν μπορεί κανείς να μειώσει τα ποσά αυτά. Δεν το ξέρω αυτό. Στην περίπτωση που τα, οι χώρες μέλη δεν δώσουν ε, ε, περισσότερα χρήματα δεν έχει νόημα ε, να πιστεύουμε ότι θα τηρήσουμε τις αυξημένες υποχρεώσεις. Μπορούμε να μειώσουμε λοιπόν και το επίπεδο των πληρωμών εγώ ήδη υπέδειξα κάποιες επιλογές. Όλα περιορίζονται φυσικά από τα περιθώρια του MFF, της ε, πολιετού συμφωνίας. Γι' αυτό όμως χρειάζεται ομοφωνία στο Συμβούλιο. Και δεν νομίζω ότι και 28 χώρες πρόκειται ποτέ γι' αυτό να διαφωνήσουν. Μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς όλες τις αναδιπλώσεις, τις μετακινήσεις, τις μεταφορές, τα ανώτατα όρια, τις ευελιξίες, αλλά ποτέ δεν θα μπορέσουμε να φτάσουμε στα 28, 29 ή 30 δις τα οποία από ό,τι φαίνεται θα χρειαστούν επιπλέον. Και μια τελευταία επιλογή και θα ήθελα και προτάσεις από πλευρά σας είναι να περιορίσουμε με κάποιο τρόπο ε, και τις πληρωμές και προς τις χώρες, ε, ε, ιδιαίτερα στον τομέα της περιφερειακής πολιτικής. Εφόσον δεν υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα, κοιτάξτε να πούμε στα κράτη-μέλη δεν μπορείτε να πάρετε επιστροφές, μπορείτε να συνεχίσετε με τα προγράμματα αυτά, αλλά εμείς χρήματα περισσότερα δεν μπορούμε να σας δώσουμε. Αυτό είναι μια επιλογή η οποία δεν θα αρέσει στα κράτη-μέλη, πρέπει όμως να τεθεί σαν <clears throat> επιλογή. Στη σύμβαση αν λέγεται ότι αν δεν πληρώσει κανείς έγκαιρα τότε θα πρέπει να πληρώσει επιτόκιο για τις καθυστερήσεις, φυσικά τα πράγματα χειροτερεύουν. Αν όμως υπάρχει η δυνατότητα να μειώσουμε κάπως τις πληρωμές, τότε θα πρέπει να πληρώσουμε πρώτα για τις ε, συμβάσεις οι οποίες είναι θα έλεγα α, κυρωτικές με την έννοια ότι αν δεν πληρώσουμε θα ε, υπάρξουν κυρώσεις εις βάρος μας, οικονομικές. Αλλιώς ε, να πούμε στα κράτη-μέλη ότι δεν θα πάρουν τα χρήματά τους πίσω. Νομίζω ότι το θέμα αυτό θα τεθεί για τα επόμενα χρόνια αρκετά συχνά. Ακόμα και τους επόμενους μήνες λέει ο κύριος Λαμασούρ, όχι μόνο τα επόμενα χρόνια. Γιατί ξέρετε ότι υπάρχει και η προεκλογική εκστρατεία για κάποιους από μας. Αν θέλεις να συμπληρώσεις. Ναι. Νομίζω ότι είναι πολύ ανησυχητικά όλα αυτά, γιατί οι ανάγκες πληρωμών για τις οποίες συζητούμε είναι πληρωμές για παλιές συμβάσεις. Ε, είναι όροι που θα πρέπει να πληρωθούν. Και κοιτώντας ε, τη γραφική παράσταση που δεν απατώμενη στη σελίδα 4 και δείχνει τις επιπλέον ανάγκες που αναμένονται για το 2014 με 711 εκατομμύριο ο Γιάν μίλησε για λίγα περισσότερα κονδύλια για την έρευνα, αλλά υπάρχουν και άλλα ενδεχομένω για το Ταμείο Απαγκοσμιοποίηση ε, ή το Ταμείο Λιλεγγύης. Και επίση κινητοποίηση του αποθεματικού για τις κατεπήγουσες έκτακτες ανάγκες. Αυτό τι δείχνει, ότι το δικό μας επιχείρημα, για το οποίο συμφωνούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, που λέει ε, ότι οι πληρωμές ε, ε, θα πρέπει να ξεπερνούν την οροφή αυτή, το πλαφόν που έχουμε βάλει. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να το τονίζουμε φέτος. Εμείς έτσι έχουμε ερμηνεύσει τη συμφωνία και ξαφνικά έχουμε βρεθεί σε μια κατάσταση όπου δεν χωράει καμία αμφιβολία. Έτσι θα πρέπει να προχωρήσουμε και έχει ξεπεράσει την οροφή και τελείως. Αναφέρονται και κάποια άλλα μέτρα, όπως και ο Γιάννη Μέλντερ αναφέρθηκε σε αυτά, πώς μπορούμε να το ξεπεράσουμε, να μειώσουμε το επίπεδο ε, ανάληψης υποχρεώσεων. Στην περιφερειακή πολιτική έχουμε δει ότι υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη που έχουν δυσκολίες στην εφαρμογή του, στην εκτέλεση δηλαδή των προγραμμάτων και των κονδυλίων που τους έχουν ε, δοθεί και έχουμε και τη ρήτρα εκπνοή, τη λεγόμενη sunset clause. Υπάρχει πολιτική βούληση να κινητοποιηθεί αυτή και να εφαρμοστεί αυτό και να αφαιρεθούν κάποια κονδύλια. Ξέρω ότι έχει γίνει, γίνει αυτό στο παρελθόν για την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, αν δεν απατώμε, έχουν υποχρεωθεί να επιστρέψουν κάποια χρήματα που δεν δαπάνησαν εγκαίρως. Αλλά τι γίνεται όταν η χώρα είναι φτωχή θα υπάρξει η πολιτική βούληση να πει φέρτε πίσω τα χρήματα ή θα έρθει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το επιβάλλει. Λυπούμεθα πάρα πολύ, πήρατε τα κονδύλια αυτά, δεν τα έχετε δαπανίσει, έχει εκπνεύσει τριετία, ε, λυπούμεθα πάρα πολύ, επιστρέφονται τα χρήματα και δεν καταβάλλεται αυτή η πληρωμή. Ξαφνικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούμε όλα τα μέτρα που έχουμε και το περιθώριο ε, έκτακτης ανάγκης για να αυξηθεί το επίπεδο των πληρωμών, αλλά και το επιχείρημα του Γιάν για τον περιορισμό των πληρωμών είναι ενδιαφέρον. Αφήστε που μπορεί και να γίνεται ήδη. Σας είπα στο προηγουμένως ότι οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις ε, έχουν πληρώσουν ε, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 300.000 ευρώ σε τόκους λόγω καθυστερημένων πληρωμών. Και αυτό ισχύει για όλους τους ιδιώτες με τους οποίους συμβαλόμεθα που είναι μη κυβερνητικέ οργανώσεις και άλλες και θα πρέπει τα κράτη-μέλη να δείξουν μια υπομονή και να περιμένουν τα χρήματα αν δεν μπορούν τα ίδια να δώσουν. Εκεί μπορούμε κάπως να καθυστερήσουμε τις πληρωμές, αλλά για κάποια κράτη-μέλη θα είναι οδυνηρό και αυτό. Ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποιες χώρες που αντιμετωπίζουν τεράστιες οικονομικές δυσχέρειες και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Merci. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ, Αν. Κύριε Γενικέ, Διευθυντά, έχετε παρατηρήσει σχόλια μετά από όλες αυτές τις ε, τοποθετήσεις. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όχι, δεν νομίζω. Η ανάλυση του κυρίου Μέλντερ είναι πάρα πολύ εμπεριστατωμένη και πλήρης για τις λύσεις. Όντως, ε, αντιμετωπίζουμε μια τεράστια δυσκολία. Διότι υπεθυμίστηκε ότι πρέπει να πληρώσουμε υποχρεώσεις του παρελθόντος και δεν έχουμε άλλη λύση. Είμαστε υποχρεωμένοι να εξοφλήσουμε αυτές τις οφειλές. Τελεία και παύλα. Ταυτόχρονα όμως, εάν θέλουμε να πούμε ότι η λύση ε, Βέβαια υπάρχει κάποια ευελιξία περιορισμένη ε, σε σχέση με τις υποχρεώσεις. Εάν η λύση λοιπόν περνάει μέσα από την ανάληψη υποχρεώσεων, πώς θα γίνει αυτό, ποιες υποχρεώσεις. Ε, η ανάληψη υποχρεώσεων αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων, ομόφωνη μάλιστα, του δημοσιονομικού πλαισίου, που ορίζει και οροφές και ανώτατα όρια. Γνωρίζουμε πολύ καλά. Τι περιμένουν τα κράτη-μέλη που απεφελούνται ως δικαιούχοι. Περιμένουν οι δαπάνες να τους καταβάλλονται. Και αυτή τη στιγμή αλλάξουμε κάτι στην ανάληψη υποχρεώσεων, θα αλλάξουμε αναγκαστικά και κάτι, όχι περιφερειακού, περιθωριακού χαρακτήρα, ε, στην ισορροπία του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου, στην πολιτική μάλιστα ισορροπία. Εάν θέλουμε να μειώσουμε την ανάληψη υποχρεώσεων, τι θα μειώσουμε, τα ποσά από ποιο τίτλο, το 1α, ένα β 2, 3, τέσσερα την την έχουμε περικόψει αρκετά. Ομολογώ ότι θα έχω πολύ μεγάλη δυσκολία να προτείνω κάτι. Ανα, ε, αναφερθούμε στην ετήσια συζήτηση για τον προπολογισμό στο Συμβούλιο. Τι βλέπει κανείς εκεί. Οι καθαροί συνεισφορείς έχουν την τάση να θέλουν να μειώνουν τα ποσά για τη συνοχή άμεση αντίδραση των ε, καθαρών ε, ε, δικαιούχων ότι θέλουν να μειώσουν τα ποσά για τη γεωργία που θίγει και για κάποιες ευαισθησίες είτε στον τίτλο 1α και τι διαπιστώνουμε ότι αλληλοεξουδετερώνονται αυτοί και τελικά οι περικοπές που γίνονται λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, σε ένα α όπου ο καθένας θεωρεί ότι έχει μεγαλύτερη ελευθερία και αυτό είναι εις βάρος της ανάπτυξης. Τα περιθώρια όμως είναι πάρα πολύ περιορισμένα. Έτσι έχουμε περιέλθει σε μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη και κατά την άποψη μου μόνος τρόπος να ξεφύγουμε είναι να ε, αντέξουμε, να κινητοποιήσουμε τα μέσα ευελιξία στο σύνολό τους και ουσιαστικά το Συμβούλιο να αναγκαστεί να δεχθεί ότι ό,τι ανάληψη υποχρεώσεων υπάρχει θα πρέπει να συνοδεύεται από την αντίστοιχη πληρωμή. Και αυτό που κάνουμε, το κάνουμε ήδη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι να επευραδύνουμε το ρυθμό της καταβολής των πληρωμών όπου μπορούμε. Οι χώρες που το έχουν λιγότερο ανάγκη αναγκάζονται να περιμένουν περισσότερο για να εξοφληθούν και ε, δίνουμε και επικεντρώνουμε την προτεραιότητά μας στις χώρες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Πάντως προσπαθούμε να ξεπεράσουμε αυτή τη δύσκολη κατάσταση που είναι υψηλές οι πληρωμές, πάντα ε, με πολύ μεγάλη συγκράτηση ε, και εν ώψη της ενδιάμεσης ε, ενδιάμεσης περίοδου. Και εκεί θα τεθεί το εξή πολιτικό ερώτημα κατά τη γνώμη μου για την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που λέει το εξή. Δεδομένης της κατάστασης που θα επικρατεί τότε, μήπως χρειάζεται να ε, επέμβουμε για τις ε, πληρωμές. Αυτό όμως είναι για πολιτική συζήτηση και θα αφορά τους επόμενους ε, βουλευτές. Ευχαριστώ κύριε Γενικέ. Ο Σαλβαδόρ Γαρίγα. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Η συζήτηση αυτή τώρα είναι ακόμα πολύ νωρί, πολύ πρόωρη, δόξα τω Θεώ, αλλά το επόμενο κοινοβούλιο, αλλά και το παρόν ακόμα, ε, τον Ιούνιο κάπως θα πρέπει να αποφανθεί για την ε, απαραίτητη ε, πρόβλεψη για τον προπολογισμό για τις πληρωμές το 2015. Από τις διάφορες λύσεις που προτείνονται, το πρώτο που θα πρέπει κανείς να σκεφτεί είναι ότι δεν θα απορροφηθούν οι πιστώσεις 2014-2020 καθόλου. Διότι όπως πολύ καλά γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα επιχειρησιακά σχέδια στην καλύτερη περίπτωση θα εγκριθούν ε, το φθινόπωρο και μάλιστα όχι αρχές φθινοπόρου. Οπότε δεν θα έχουμε ε, μεγάλες αναλήψεις υποχρεώσεων εκεί και για το υπόλοιπο προς εκαθάριση που έχει συσσωρευτεί από την προηγούμενη περίοδο. Η ιδέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως μας την πρότεινε ο κύριος Λεβαντόφσκι, ε, έχει ως εξής. Το πρώτο του χρονοδιάγραμμα πληρωμών, σε αυτό ουσιαστικά βασιζόταν ότι οι υφιστάμενες πληρωμές από το 2014 θα καλύψουν την προηγούμενη περίοδο. Τώρα θα χρειαστούμε και μια αξιολόγηση και από την άλλη, από τις διάφορες λύσεις που προτείνονται και που πρότεινε ο συνάδελφος Μόλντερ, βλέπω πολλές δυσκολίες. Πρώτον, αυτές οι αποφάσεις είναι πολιτικές και εξ όσων εγώ κατανοώ, αυτό αφορά τα δύο σκέλη του, δημοσιονομικής αρχής. Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία και κοινοβούλιο ανάλογα με τις πολιτικές ομάδες και την εκάστοτε εθνικότητα των παρόντων λαμβάνει αποφάσεις για το εάν και κατά πόσο μπορεί να γίνει μείωση στις πιστώσεις ανάληψη υποχρεώσεων. Αυτή θα φαινόταν η πιο λογική λύση. Θυμάστε όμως πολύ καλά ότι έχουμε κάνει αυτή τη συζήτηση προηγούμενα έτη εδώ στην Επιτροπή Προλογισμών ακριβώς επειδή αυξάνεται συνεχώς το προσεκαθάριση υπόλοιπο, μήπως χρειάζεται και είναι σκόπιμο να μειωθούν οι δαπάνες για ε, πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων. Και η τελική μας ε, απόφαση ποια ήταν το συμπέρασμα, ότι είναι πολιτική βούληση αυτή που εκφράζεται από το Κοινοβούλιο στην ανάληψη υποχρεώσεων και έτσι καταδεικνύουμε και τις προτεραιότητές μας. Βέβαια τώρα η μείωση των πιστώσεων ανάληψη υποχρεώσεων θα σημάνει ότι καλείται το Κοινοβούλιο να αναθεωρήσει τις ίδιες του τις πολιτικές προτεραιότητες. Αυτό είναι θέμα του επομένου Κοινοβουλίου και της επομένης θητείας. Αλλά θα έρθουμε αντιμέτωποι με αυτή την κατάσταση. Από την άλλη, επίση το Ταμείο είναι μείον στα μέσα ευελιξία. Ούτε φαίνεται πάρα πολύ αναγκαίο να τα εξαντλήσουμε αυτά τα κονδύλια, γιατί θα χρειαστεί μετά το 2015 να τα βρούμε ξανά όταν θα έχει επιταχυνθεί ο κύκλος τη της οικονομίας. Ε, το πιο λογικό νομίζω το είπε ο κύριος Γενικός Διευθυντής ότι κανονικά θα πρέπει να περιμένουμε την διάμεση αναθεώρηση των δημοσιονομικών προοπτικών όπου θα χρειαστεί οπωσδήποτε να αυξηθούν οι οροφές για τις πληρωμές. Αυτά το γνωρίζουμε όλοι. θα πρέπει να υπάρξει σημαντική αύξηση και πραγματική αναθεώρηση των δημοσιονομικών προοπτικών. Αυτό όμως για να γίνει θα πρέπει το οικονομικό περιβάλλον να είναι πολύ διαφορετικό από το σημερινό. Με την ε, δημοσιονομική εξηγίαση των κρατών μελών να έχει δώσει τη θέση της ε, σε ανάπτυξη με συλλογή φόρων στα κράτη-μέλη. Σήμερα μια τέτοια συζήτηση στα κράτη-μέλη είναι αδιανόητη. Για νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ένα ημερολόγιο για τις πληρωμές και ένα χρονοδιάγραμμα αρκετά πιεσμένο. Αυτά για το 2014, για το 2015 θα συζητήσουμε για την εκτέλεση των νέων δημοσιονομικών προοπτικών και για τις οροφές των πλήρωμων. Προς στιγμή δεν, νομίζω, δεν πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε τίποτα παραπάνω. Καλό είναι όμως να γνωρίζουμε την κατάσταση, να αρχίζουμε να προειδοποιούμε τις πολιτικές ομάδες και τα κράτη-μέλη για το ποια είναι η πραγματική κατάσταση των οικονομικών μας δεν μπορούμε όμως να κάνουμε τίποτα παραπάνω αυτή τη στιγμή, απλώς να ε, κρούσουμε τον κόδωνα του κινδύνου και να πούμε το 2015 θα τα βρούμε μπροστά μας αυτά τα προβλήματα. Ευχαριστώ Σαλβαδόρ. Είναι σοβαρό το πρόβλημα. Έλεγα προηγουμένως ότι μπαίνουμε σε προεκλογική εκστρατεία για την ανανέωση της Ευρωβουλής και σαν μέλη της Επιτροπής Προϋπολογισμών όταν παίρνουμε μέρος στην προεκλογική εκστρατεία έχουμε το καθήκον να ενημερώνουμε τα πολιτικά μας κόμματα, τους συμπολίτε μας, γιατί στην παρούσα στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει τα μέσα για να ασκήσει τις πολιτικές της και τους στόχους που θέτει το Συμβούλιο και ότι στα πλαίσια της επόμενης κοινοβουλευτικής περίοδου πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα συμπεράσματα. Κάποιοι θα πούν ότι θα πρέπει να μειωθούν οι, οι φιλοδοξίες, άλλοι τα μέσα, άλλοι και τα δύο, άλλοι να βρούμε νέους ιδίους πόρους, γιατί θα τεθεί σε λειτουργία και η ομάδα υψηλής επαφής για τη μεταρρύθμιση της χρηματοδότησης του προϋπολογισμού. Νομίζω πάντως ότι στα πλαίσια της προσπάθειας που γίνεται έχουμε κάποιους αριθμούς που θα μας επιτρέψουν να πούμε το τι έχουμε στη διάθεσή μας και ποια είναι τα ράλλα, ποια είναι τα υπόλοιπα προς εκαθάριση, δηλαδή τα σορευμένα χρέη τα οποία θα πρέπει να πληρωθούν και με τα οποία οι διάδοχοί μας θα πρέπει να διαχειριστούν τον κοινοτικό προϋπολογισμό με όλες τις δυσκολίες οι οποίες ε, ήρθαν στην επιφάνεια από το απόγευμα στα πλαίσια του Monitoring Group και τη συζήτηση για τα υπόλοιπα προς εκαθάριση. Αυτή είναι η προσωπική μου ε, θα έλεγα αίσθηση και αυτό θα κάνω κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Δεν ξέρω αν οι, οι θέλουν να πούν κάτι άλλο. Δεν θέλει κάποιος άλλος το λόγο. Σας ευχαριστώ όλους. Εξαντλήσαμε την ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας της Επιτροπής μας για σήμερα. Τέλος λοιπόν των εργασιών, μέχρι αύριο το πρωί, 9η πρωινή, θα ξεκινήσουμε με τις ψηφοφορίες. Αλλά όμως θα ήθελα να μείνουν εδώ οι συντονιστές, γιατί ταυτόχρονα θα γίνει η συνάντηση των συντονιστών και θα ζητήσω από τους διερμηνείς που ανταποκρίνονται στους παρόντες εισηγητές να παραμείνουν στην αίθουσα. Υποτίθεται ότι είναι ήδη ενημερωμένοι γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά, ισπανικά, λόγω του γνωστού Σαλβαδόρ. Άλτα δεν είναι εδώ, οπότε δεν θα χρειαστούμε την πορτοκαλική. Λοιπόν, οι υπόλοιποι διερμηνείς μπορούν να αποχωρήσουν. Ε, πρέπει να αποχωρήσουν επίσης και όσοι δεν συμμετέχουν στη συνάντηση των συντονιστών και να έρθουν οι απόντες συντονιστές.